να αναπτύξουν μια επαρκή συνεργασία. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω για την δική μου στεναρή πεποίθηση όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα και τη δέσμευση. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπαρνιέ. Ε, κύριε συνάδελφε, έχει κλείσει η συζήτηση και θα γίνει η ψηφοφορία αύριο στις 12 για το θέμα αυτών των τυχερών παιχνιδιών online. Τώρα θα συζητήσουμε για τη μελισσοκομία. Υγεία των και Υγεία των μελισσών και μελισσοκομικό τομέα. Ο εισήγητή έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Νταλή, εγώ μιλάω κυρίως για την υγεία, στην έκθεσή μου για την υγεία των μελισσών, αλλά μιλάω και για άλλα σημαντικά θέματα που αποτελούν πρόκληση για μας ε, και που αφορούν τον κλάδο αυτό. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσίασε μια θαυμάσια ανακοίνωση και η έκθεσή μου βασίστηκε σε αυτό το έγγραφο. Προσπάθησε να, το... να ξεκινήσει από εκεί και να πάει ακόμη πιο πέρα. Σε αυτή την έκθεση κάνουμε διάφορες προτάσεις, τις οποίες ελπίζω να λάβει υπόψη η Κομισιόν, τα κράτη-μέλη και ο κλάδος στα κράτη-μέλη. Το διακύβευμα δεν είναι μόνο η παραγωγή μελιού αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι πολύ σημαντική η επικονίαση για όλο το γεωργικό κλάδο και για την διατήρηση της βιοπικιλότητας. Σκεφτείτε ότι το 85% των καλλιεργειών είναι εφικτό μόνο χάρη στην δραστηριότητα των μελισσών που είναι οι βασικοί επικονιαστές. Αλλιώς δεν θα υπήρχε γεωργία. Επομένως η μελισσοκομεία έχει πολύ πιο ευρεία λειτουργία ε, στο εσωτερικό της γεωργίας. Ε, επομένως θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτό τον ε, κλάδο με κοινοτικά κονδύλια, με ενωσιακά κονδύλια. Εδώ και δεκαετίες, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είχαμε αρκετά φάρμακα για τις μέλισσες. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται να παράγουν νέα φάρμακα για τον κλάδο της μελισσοκομείας. Και ο μελισσοκομικός κλάδος από μόνος του δεν έχει αρκετά κονδύλια για να χρηματοδοτήσει την δημιουργία νέων φαρμάκων. Εδώ και χρόνια σέρνουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν δεν παρέμβουμε εμείς με ενωσιακά κονδύλια, αυτή η κρίση η οποία πλήττει τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μελισσοκομικό τομέα δεν θα ξεπεραστεί. Ένα άλλο πρόβλημα σοβαρό είναι ότι αυτός ο κλάδος δεν είναι αρκετά οργανωμένος. Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα, αξιόπιστα, δεν υπάρχουν μελέτες για τον αριθμό των μελισσοκόμων, για τον αριθμό των κυψελών, για το, τη θνησιμότητα των μελισσών και πού οφείλεται. Επομένως, πρέπει να έχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αξιόπιστα δεδομένα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η επαγγελματική ενημέρωση των μελισσοκόμων. Θα ήταν πολύ σημαντικό στα κράτη-μέλη να οργανωθεί ένα είδος επαγγελματικής κατάρτιση υποχρεωτικής για του μελισσοκόμους. Ένα άλλο θέμα προσυζήτηση είναι η επιρροή των φυτοϊγειονομικών προϊόντων στη θνησιμότητα των μελισσών. Υπάρχουν κάποιοι γεωργοί οι οποίοι θέλουν να λύσουν το πρόβλημα ε, χύνοντας ε, ε, φυτοφάρμακα. Εγώ δεν συμφωνώ. Θα πρέπει να μειώσουμε τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Και λυπάμαι που ορισμένοι δεν επέτρεψαν να μπει σε αυτή την έκθεση ο αριθμός αυτών των φυτοϊγειονομικών προϊόντων που είναι επικίνδυνα και τοξικά και ποια είναι τα βασικά ενεργά στατικά αυτών των προϊόντων που μπορούν να σκοτώσουν τις μέλισσες και μπορούν να αντικατασταθούν όμως από προϊόντα λιγότερο τοξικά. Παραδείγματο χάρη μιλάω για τα νοικοτινοειδή, αυτά τα ενεργά, ε, τις ενεργές ουσίες που θα πρέπει να αντικατασταθούν από πιο ε, οικολογικά προϊόντα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν νέες ενεργές, ναι, νέες ενεργές ουσίες στα φυτοφάρμακα. Θέλω επίσης, Κομισιόν, να τροποποιήσετε την οδηγία για το μέλι, γιατί σε αυτή την οδηγία δεν ε, αναφέρονται επαρκώς οι, τα στοιχεία και οι παράγοντες ε, ποιότητας του μελιού. Όταν γίνεται υπάρχουν μέλια από μιμήσεις, ας πούμε μέλια μαϊμούδες κτλ. Εμείς δεν έχουμε κανένα εργαλείο για να παρέμβουμε. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για τα κράτη-μέλη που εξάγουν ε, τα προϊόντα τους. Επίση, οι γάματα φόμικρον, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Και εδώ γίνονται πολλέ συζητήσει. Είναι επικίνδυνε αυτέ οι Δεν είναι. Σε ποιο βαθμό είναι. Εγώ καλώ την Επιτροπή να ξεκινήσει ε, και να ζητήσει μια αντικειμενική επιστημονική μελέτη, γιατί αυτό δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα επιστημονικό. Δεν έχουμε όμως ε, στη διάθεσή μας επιστημονικά στοιχεία και μελέτες. Ό,τι αφορά τα αντιβιωτικά, θα ήθελα να σας ζητήσω, Επίτροπε, να ρυθμίσετε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη για τα κρέατα. Υπάρχουν ε, ανώτατα όρια καταλήπων αντιβιωτικών. Ε, για το μέλι δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Καλό θα ήταν να έχουμε λοιπόν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τέτοια ανώτατα όρια. Επίσης, υπόθηκε ότι αν ε, εξαλειφθούν οι μέλισσες από τον πλανήτη, μετά από τέσσερα χρόνια θα εξαλειφθεί η ανθρωπότητα. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η επίπτωση της μελισσοκομείας για την ανθρωπότητα και τη διατήρηση της βιοπικιλότητας. Ε, γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτό που είπε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, γιατί αυτός το είπε αυτό. Έχουμε πάρα πολλές αιτήσει ε, για το μικρόφωνο. Προσοχή. Όπως υπόθηκε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα από τον προηγούμενο μιλητή, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και πολλά διακυβεύονται. Ε, ο Αϊνστάιν ήξερε πόσο σημαντικό είναι το θέμα των μελισσών και της μελισσοκομίας και η παράθεση αυτή από τον συνάδελφο είναι σημαντική. Ε, το 35% των μελισσών ε, εξαρτώνται από την επικονίαση. Αν εξαλειφθούν οι μέλισσες, όπως είπε και ο Αϊνστάιν, θα εξαλειφθούν πολλά είδη. Ε, κάτι που κάνουμε ε, επιτυχώς στην ε, Ιρλανδία είναι ότι προστατεύουμε τις μέλισσές μας. η καθαρότητα διαφόρων ειδών πρέπει να προστατευθεί. αυτό το θέμα είναι τεράστιο, είναι μείζον. Και για την οικονομία ακόμα. Αν αυξήσουμε την την πρόσληψη μελιού στην καθημερινή μας διέτα θα βελτιώσουμε και την υγεία μας. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε το γεγονό ότι η υγεία των μελισσών σε εποχέ ε, κρίσης προφανώς δεν μπορεί να προσλάβει αυτή την σημασία που της αξίζει είναι προφανές, αλλά είναι εσφαλμένο. Ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε πει ότι η ανθρωπότητα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει τέσσερα χρόνια με τι μελισσές. Η υγεία των μελισσών αφορά την γεωργία, την παραγωγή τροφίμων, τη διατήρηση της βιοπικιλότητα και τέλος την ίδια μας τη ζωή εάν εξαλειφθούν οι μέλισσες και αναφέρουμε σε ορισμένες περιοχές της Αυστρίας όπου το ποσοστό αυτό είναι 30%. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνουν έρευνες ε, για το φαινόμενο αυτό, αλλά δεν θα πρέπει αυτό να παραμείνει το μόνο βήμα. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένη καθοδήγηση μέσω ενισχύσεων στη γεωργία και συγκεκριμένες διαδικασίες όσον αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα γιατί η σύγχρονη γεωργία πραγματικά ε, είναι υπεύθυνη. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ενίσχυση για την έρευνα, για βελτίωση της υγείας των μελισσών, για πρόληψη και για αποτελεσματική τυποποίηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων στις χώρες μέλη και για εναλλακτικές δυνατότητες για ε, προσταχημικά ε, παρασιτοκτόνα, δηλαδή μέσω βιολογικών. Ευχαριστούμε πολύ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 Γι' αυτό εμείς ε, θέλουμε ένα εναλλακτικό ψήφισμα. Τα νεονικοτοειδή θα πρέπει να αποσυρθούν τώρα από την αγορά γιατί λέγεται ότι διαδραματίζουν ένα αρνητικό ρόλο. Επίσης οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Εδώ υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι στη βάση της αρχής της πρόληψης θα πρέπει να μην υπάρχουν γενετικά, γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Χρειαζόμαστε περισσότερη αμυψη και λιγότερες μονοκαλλιέργειες. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να προσεγγιστούν αποτελεσματικά για να επιληθεί το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Το, το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκής Ένωση το Σεπτέμβριο απεφάνθη ότι όλα τα ε, μπολάκια μέλη θα πρέπει να φέρουν ετικέτα που να λέει ότι εμπεριέχεται βασιλικός ε, γύρι μέσα στο, ε, στο μέλι. συγγνώμη, ένα πεντάχρονο μπορεί να σας το πει αυτό. Δηλαδή είναι να βάζουμε πάνω στα φιστίκια μία ετικέτα και να λέμε μπορεί να περιέχονται ίχνη από φιστίκια ή από ξηρούς καρπούς. Ε, όταν μιλάμε για τις ασθένειες, ε, για την ε, βαροϊκή νόσο, για την μετατόπιση των μελισσιών και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε πόσα προβλήματα υπάρχουν στον τομέα αυτό, αλλά δεν έχει καμία σχέση τώρα με τις ετικέτες. και ούτως ή άλλως οι δικαστέ δεν έχουν καμία θέση να αποφασίσουν γι' αυτό. Εμείς οι νομοθέτε εδώ θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να αναφέρουν οι ετικέτε. Δηλαδή τι είναι στο αρχηγείο τους ε, στο Λουξεμβούργο και αποφάσισαν να πούμε τους ήρθε επιφύτηση και είπαν ότι μεγάλη σοφία ότι ένα κουτί με πιστίκια περιέχει ξερούς καρπούς. Ο κύριος Φερέιρα τώρα ευχαριστώ. Ε, η συνεχής αποδυνάμωση των απικιών των μελισσών ε, είναι ένα πολύ ανησυχητικό πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια ε, ουσιαστική αποτελεσματική λύση. Αυτή ο, επηρεάζει όχι μόνο τις ε, ημέρες αλλά και τις άγριες μέλισσες που κάνουν την επικονίαση και συνειδητοποιούμε πόσο επηρεάζει αυτό το φαινόμενο και τη γεωργία και γενικότερα τα οικοσυστήματα. Δεν μπορούμε παρά να θέσουμε υπό αμφισβήτηση τι καλλιεργητικέ ε, μεθόδου. Επικρατεί η μονοκαλλιέργεια. Ε, Επίση, ολένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται βιοχημικέ ουσίε, ζυζανιοκτώνα, διαδίδονται οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Δεν υπάρχει καμία εφαρμογή τη αρχή τη πρόληψη. Ε, θα πρέπει να ανεληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα, να καταργηθούν ε, ε, διάφορα προϊόντα, αλλά πέραν αυτού χρειάζεται και επιστημονική στήριξη από τους γεωργικούς, ε, αλλά και μέτρα ουσίας. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι καλλιεργητικές ε, πρακτικές, καθώς και οι πολιτικές που τους υποστηρίζουν. Η μεταρρύθμιση κοινή γεωργικής πολιτικής θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την τροποποίηση. Αλλά οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν οδεύουν προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε η κυρία Πατρέων τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή και τους Σκιώδης ε, για την καλή δουλειά που έκανα. Θα ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που παρά τις προσπάθειές μου δεν συμπεριλήφθηκε μέσα στο κείμενο. Ε, η δήλωση σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης υποειδών εκτός του φυσικού τους περιβάλλοντος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ε, και καλούνται αυτά τα έντομα να επιβιώσουν σε συνθήκες που όμως δεν ε, ταιριάζουν με το φυσικό τους περιβάλλον. Ε, δηλαδή για την παραγωγή μελιού υποσκάπτουμε την άμυνα παραδείγματος χάρη των εντόμων και θέτουμε σε κίνδυνο τις ζωές τους, εισάγουμε εξωτικές ασθένειες και χρησιμοποιούνται εγχώρια ή υποείδη χωρίς να είναι ενημερωμένοι οι ε, θα πρέπει να σταματήσει αυτή η πρακτική άμεσα διότι πλήττει τους πάντες. Σας ευχαριστούμε. κυρία Μέρκη στην επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Εγώ υποστηρίζω το εναλλακτικό ψήφισμα που θα ψηφιστεί αύριο. Εξηγήσαμε εξηγούμε την γονιμότητα στα παιδιά, τη σεξουαλικότητα. Ξεκινάμε με τα... Με μεταφορές, ας πούμε, βασίζονται στις ε, μέλισσες. αν πεθάνουν οι μέλισσες, δεν θα μπορούμε καν να χρησιμοποιούμε αυτά τα παραδείγματα. Ε, θα χάσουμε και πολλά προϊόντα, όμως. Νομίζω ότι αλλάζουμε άρδιν τη φύση έτσι. Και το κάνουμε μάλιστα με λάθος τρόπο. Δηλαδή, επιτρέπουμε τους ε, γεωργού, στους γεωργούς να χρησιμοποιούν πάρα πολλά ε, φυτοφάρμακα, τους επιτρέπουμε εντατική γεωργία, μονοκαλλιέργειες. Είναι λάθος ο τρόπος προσεγγίζουμε την ε, γεωργία. Για να ξαναδούμε λιγάκι τη βιολογία μας, το μάθημα βιολογίας, για να ξαναδούμε ε, πώς αναπαράγονται οι μέλισσες και τα πουλιά. Bees, like Όπως οι Ρωμά και οι μέλισσες έχουν ελεύθερο πνεύμα. Δεν τους ενδιαφέρει ε, από πού προέρχεται η γύρι που συλλέγουν. Ε, για, για, ρωτήστε για ρωτήστε κάποιον ε, που είναι σε ένα λεωφορείο ε, από πού προέρχεται αυτή η γύρι. Ε, δεν έχει ιδέα. Ε, αυτό που ισχύει για τους ε, εμπόρους, τους Ρωμά, ισχύει και για τους ε, μελισσοκόμους. Ε, νομίζω ότι δεν μπορούν να να... αυτά που τους επιβάλλουν δεν μπορούν να τα σεβαστούν ε, οι μελισσοκόμοι και κλείνουν τα μαγαζιά τους, κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρο και ευχαριστώ τον εισηγητή. Θα προτιμούσα η έκθεση αυτή να είναι για μέλισσες και βασιλικές μέλισσες. Ε, πριν ε, κανείς καταλήξει κάποια συμπεράσματα για τις αίτιες του προβλήματος, η έκθεση ε, μιλά για έλλειψη σε σχέση με θέματα που αφορούν την απώλεια κυψελών και χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα που να μας παράσχει πληροφορίες επί των οποίων να βασιστούμε. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Η βασική ε, η ιδέα ότι τα παρασυντεκτόνα δημιουργούν το πρόβλημα θα πρέπει να εξεταστεί αλλά ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει μια δεν θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση με νέα παρασετοκτόνα. Ε, θα πρέπει οι κότοποι όλων των ε, εντόμων να ε, γίνουν σεβαστοί. Εγώ είχα τέτοιες καλλιέργειες και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μακίνες. Τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ντάλι, τον Επίτροπο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι έχουν γίνει πολλές συζητήσεις φέτος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη μελισσοκομεία. Δείχνει, αυτό δείχνει ότι αυτή η ανακοίνωση υπήρξε ένα εργαλείο για την ενίσχυση μιας καλύτερης συνεννόησης στο θέμα αυτό. Η αρχική μας αξιολόγηση παραμένει έγκυρη. Η υγεία των μελισσών επηρεάζεται εντόνως από διάφορους παραμέτρους, ενώ σήμερα η επιστήμη δεν έχει ακόμα καθορίσει τις ακριβείς αιτίες ή την έκταση της απώλειας των μελισσών. Επιτρέψατε μου να εκφράσω εδώ την εκτίμησή μου για την εξαίρετη εργασία της εισηγήτριας της κυρίας Σταπάκη, η οποία πραγματικά συνέταξε μια ισορροπημένη έκθεση σε αυτό το πολύ σύνθετο θέμα. Ε, ε, δυστυχώς συμφωνούμε ότι ε, δεν υπάρχουν εύκολες ε, ή ενιαίες ε, λύσεις. Ωστόσο είναι ξεκάθαρτο ότι οι ερευνητικές προσπάθειες θα πρέπει να συνεχίσουν και θα πρέπει να δώσουμε προσοχή στην επιλογή μελλοντικών ερευνητικών προγραμμάτων γιατί θα πρέπει να εντοπίσουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία ασκούν την περισσότερη επιρροή. Η Επιτροπή ήδη εντόπισε 7 τομείς δράση όπως είναι ο ορισμός ενός, η ενός νέου εργαστηρίου για την υγεία των μελισσών και η αύξηση των κονδυλίων για την ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων. Ε, θα ήθελα πραγματικά να εκτιμήσω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Η έκθεση του Κοινοβουλίου ασφαλώ μα δίνει τροφή για σκέψη σε σχέση με τα θέματα αυτά και για πολλά άλλα επιπρόσθετα σημεία. Και μπορώ να εξασφαλίσω ταξότιμα μέλη ότι θα εξετάσουμε όλε σα τι υποδείξει ε, εκ του σύνεγγυ. Και είμαι πεπισμένο ότι η δράση μα θα μα βάλει σε μια καλύτερη θέση για να αποφασίσουμε για τι ευέλθιστε δράσει και στρατηγικέ. Θα ήθελα ωστόσο να σα υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή έχει περιορισμένου ε, πόρου και εργαλεία. Οι χώρε, μέλη και ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επίσης να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επένδυση περαιτέρω προσπαθειών στην ανάπτυξη και πρόθεση στην αγορά κτηνιατρικών φαρμάκων. Ε, ε, επίσης θα πρέπει να προωθούν οι βέλτιστες σε μελισσοκομικές πρακτικές ώστε να υπάρξει ο διάλογος μεταξύ παραγωγών ε, σπόρων και μελισσοκόμων, ούτω ώστε να υπάρξει ανταλλαγή των ε, σωστών πληροφοριών και ενημέρωση των μελισσοκόμων. Θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την αξιόλογη έκθεση του Κοινοβουλίου και θα ήθελα να πω ότι αναμένω με ενδιαφέρον τη συνέχιση ε, της, των εξελίξεων και της μίας περτέρου προόδου για αυτό το σημαντικό θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η συζήτηση έχει περαταθεί και η ψηφοφορία, όπως και για τα άλλα θέματα, θα λάβει χώρα αύριο στις 12. Ε, Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη